Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Responsibility for this uh, joint meeting. Καλημέρα σας. Με πολύ χαρά κυρίσω την έναρξη αυτής της κοινή μας συνεδρίασης ε, από κοινού με την ε, ΙΜΚΟ. Είναι εδώ η Βίκη Φόρντ. Έχουμε μεγάλη εμπειρία. Ε, έχουμε μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους ε, συνεδριάσεις και πολύ καλής ε, συνεργασίας ε, για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Πρόκειται για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Τώρα πρέπει να συνεργαστούμε για τη σχετική νομοθεσία, αλλά είναι βάση του κανόνα 55. Είμαστε δύο αρμόδιες επιτροπές για το θέμα αυτό, οπότε θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους και από τις δύο επιτροπές. Να σας συγχαρώ, κυρία Φόρντ, γιατί έχετε επανεκλεγεί πρόεδρος. Οπότε και οι δύο πρόεδροι ε, είναι ίδιοι με πιο πριν, δεν ξέρω τώρα το δικό σας προεδρείο. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Εμείς έχουμε μία μικρή διαφορά ε, στους αντιπροέδρους. η πρόεδρος και οι τρεις πρώτοι αντιπρόεδροι είναι όλες γυναίκες και είμαστε πάρα πολύ ε, περήφανοι γι' αυτό γιατί σε άλλες ε, ε επιτροπές ε, είναι ε, άντρες. Είναι η κυρία Κοράτσα Μπίλντ πρώτη αντιπρόεδρος και η κυρία Στάινερ μετά. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Η φίλη μου η Βίκη θα είναι προ, πρόεδρος της δεύτερης, ε, του δεύτερου τμήματος της συνεδρίασής μας. Βλέπετε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε καμία αντίρρηση, μπορούμε να την εγκρίνουμε. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να θέλει να, κανένα να θέλει να αλλάξει την ημερήσια διάταξη. Τώρα, ως προς τις ανακοινώσεις μου. Έχουμε διερμηνία προς όλες τις γλώσσες. Αυτό είναι καταπληκτικά νέα. Τώρα, ως προς τη διαδικασία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ καλή συνεργασία, κυρίως δε την ε, κυρία Φόρντ και τους ε, συνεισηγητές ε, Βίρκουνερ και Ζουβά για την προετοιμασία αυτής της συνεδρίασης. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρούμε χρόνο για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις εργασίες μας. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω σε όλους ότι η έκθεση αυτή θα συζητηθεί και θα εγκριθεί κατά τις κοινέ συνεδριάσεις των ε, ε, επιτροπών μας. Θα υπάρχει μια ξεχωριστή μερίσια διάταξη για κάθε μία από τις ε, συνεδριάσεις μας αυτές τις κοινέ. Και η Προεδρία θα είναι επίσης κοινή. Και οι δύο Πρόεδροι θα ενημερώνουν κάθε φορά τι έχει αποφασιστεί στις κοινέ συνεδριάσεις. Σε συμφωνία βέβαια με τους δύο συνεισηγητές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι συνεισηγητές σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις. Το θέμα μας είναι επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά. Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ευρώπη. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων βάσει του κανόνα 55 έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Δεν έχουμε έγγραφο ακόμα, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας, γιατί όπως είπα έχουμε δύο συνεισηγητές και θα ήθελα να ζητήσω από τους συνεισηγητές μας να πάρουν το λόγο, πέντε λεπτά έκαστος, και μετά να ζητήσω από τους σκιώδεις εισηγητές να πάρουν το λόγο και θα δώσω και την ε, προεδρία στην ε, φίλη μου Δίκη για το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα εισαγωγικά σχόλια και των δύο συνεισηγητών. Δεν ξέρω, κυρία Συμπρόεδρε, αν θέλετε να πει κάτι. Όχι, νομίζω ότι θα ήθελα να πω ότι θα ανοίξω τον κατάλογο των ομιλητών για όσους δεν είναι σκιώδεις. Οπότε παρακαλώ πείτε μου αν θέλετε να πάρετε το λόγο γιατί εγώ θα είμαι πρόεδρος στο δεύτερο τμήμα της ε, συζήτησης. Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Ευχαριστούμε. Ένα. Η κυρία Βίρκουνε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Έχουμε ξεκινήσει με τον συνάδελφό μου, τον Φιλίπ Ζουβά, την εκπόνηση της κοινή έκθεσης αυτής ε, για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τη δική σας άποψη για το τι θέματα θα έπρεπε κατά την άποψή σας να περιληφθούν. Νομίζω ότι καλό είναι να αναφέρουμε κάποιες από τις πτυχές που θα έπρεπε να απασχολήσουν την Επιτροπή ίτρε. Πρώτα απ' όλα οι αγορές στον τομέα αυτό αναπτύσσονται τάχιστα και είναι παγκόσμιες που σημαίνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες προσφέρουν ένα νέο φόρουμ για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Συχνά είναι διευκολυντές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρουν ε, μεγάλη επιλογή στους καταναλωτές και Ανταγωνισμός προς τις τιμές. Γνωρίζουμε ότι επιγραμμικές πλατφόρμες δημιουργούν επίσης νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και μοντέλα. Για παράδειγμα, ΜΜΕ, οι οποίες μπορούν να ωφεληθούν από τις πλατφόρμες που προσφέρουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές χωρίς επενδύσεις σε ε, ακριβές υποδομές. Κάποιες επιγραμμικές πλατφόρμες επίσης ε, εργάζονται στο πλαίσιο της ε, συνεργατικής οικονομίας, και οικονομίας. Υπάρχουν όμω και προκλήσεις. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό μένα, γνωρίζουμε όμως αυτή τη στιγμή ότι το μερίδιο ε, της κεφαλοποίησης αγοράς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ χαμηλό. Έχουμε λίγες ιστορίες επιτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα θέλαμε περισσότερες. Γνωρίζουμε ότι περισσότεροι ε, πρωταγωνιστές είναι αμερικανικής ε, καταγωγής προέλευσης. Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη των επιγραμμικών πλατφορμών στην Ευρώπη και να τονίσουμε την, ε, την ικανότητά τους για παγκόσμιο ανταγωνισμό, γιατί αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας εν γέννη στην Ευρώπη στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να έρθουν τα εμπόδια τα οποία περιπλέκουν ε, την ομαλή λειτουργία των πλατφορμών διασυνοριακά και διαταράσσουν και την ε, λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Μια από τις βασικές προτεραιότητες οι ε, άξονες ή για να σταθεί σε επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις νοφείς είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των επιγραμμικών πλατφόρμων στην Ευρώπη. Η Ευρώπη επίσης πρέπει να παρέχει ένα καινοτόμο φιλολογικό περιβάλλον, να προωθεί την έρευνα στι τεχνολογική στην ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι σημαντικό για νέε ιδέες, για την καινοτομία. Επίσης, υποδομές θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, να εξυγχρονιστούν. Ψήλης ταχύτητα διαδίκτυο είναι σημαντικό για τη χρήση των επιγραμμικών ε, υπηρεσιών. Αν δει κανεί προσεκτικά την νομοθεσία, τουλάχιστον εγώ ε, είδα ε, κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε στον επιγραμμικό και μη επιγραμμικό κόσμο. Οι κρίσιμε υπηρεσίε και επιχειρήσει θα πρέπει να έχουν ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού ε, επιγραμμικά και μη. Το να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε δεν επιτρέπει τον δίκαιο ανταγωνισμό. Με τις νέες τεχνολογίες τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και νέες προκλήσεις. Και κάτι που φαίνεται να απασχολεί τα μάλα στο πλαίσιο της συζήτησης για τις επιγραμμικές ε, πλατφόρμες είναι η ε, ευθύνη και οι υποχρεώσεις ε, των δημοσιολαβητών. Θα δημοσιεύσει σχετικέ κατευθυντήριε γραμμέ τη Κομισιόν. Είναι σημαντικό ότι οι επιγραμμικέ πλατφόρμε αναλάβουν περισσότερη ευθύνη οι ίδιε. Θα πρέπει δηλαδή κατά του ε, μη ενδεδειγμένου περιεχομένου να λάβουν μόνοι, δράση επίσης και είναι μια δύσκολη μάχη. Αυτή είναι η εισαγωγική μου ε, ομιλία. Νομίζω ότι στην Ευρώπη αυτό πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί ένα ισοτιμό πεδίο ανταγωνισμού για τις επιγραμμικές πλατφόρμες στην Ευρώπη και αυτό το στο περιβάλλον που θα προωθεί τις επενδύσεις, να ε, τονώνει την καινοτομία στην Ευρώπη, διότι θέλουμε να είμαστε στις επιγραμμικές πλατφόρμες ε, επίσης στην κορυφή. Προσβλέπω στις δικές σας συνεισφορές και προσβλέπω επίσης και σε μια πολύ οικοδομική συνεργασία με στους τους κοιόδης εισηγητές μαζί με τον συνάδελφο, με τον κύριο Ζιβάν, προβλέπουμε να έχουμε την πρώτη συνεδρία των συντονιστών στο Στρασβούργο στην ε, Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Εκεί θα έχουμε την πρώτη δυνατότητα να συζητήσουμε, μετά από καμιά δύο εβδομάδες δηλαδή, και θα επεξεργαστούμε το σχέδιο έκθεσης 28 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία και θα σταλεί τότε για μετάφραση το κείμενο. Άρα όλο τον επόμενο μήνα θα συνεργαστούμε στενά με τον συνάδελφό μου από την Επιτροπή τον κύριο Ζιβά και με τα χαρά τώρα περιμένω να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος και τώρα συνεισηγητά κύριε Ζουβά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι πρέπει να μιλάμε για ψηφιακή επανάσταση. Και το σύμπαν αυτό δεν είναι απλώς ένας χώρος ε, συναλλαγών όπως φαντάζομασταν στο παρελθόν. Είναι ε, ένας νέος χώρος και ένα νέο κέντρο εξουσίας πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής όπου οι πλατφόρμες παίζουν σημαντικό ρόλο. Πολύ σαφώς. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε κάποια ερωτήματα, ειδικά το ερώτημα που έθεσε η συνάδελφος, η κυρία Βυρκάινεν, ότι δεν υπάρχει Ευρωπαίος πρωταθλητής ή ελάχιστοι Ευρωπαίοι πρωταθλητές ε, στις πλατφόρμες, εκτός από λίγα παραδείγματα που στην πραγματικότητα καθοδηγήθηκαν από την απουσία κανόνων παρά από την παρουσία κανόνων. Θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε σήμερα τι γίνεται με αυτή την πλατφορμοποίηση της οικονομίας ε, και τα επιχειρηματικά μοντέλα. Ε, η δημόσια ρύθμιση, οι δημόσιοι κανόνες είναι κατάλληλοι. Ε, το δίκαιό μας ε, είναι σε θέση να απαντήσει στα, στις προκλήσεις του, της επανάστασης αυτής, το κοινωνικό, το φορολογικό, το επιχειρησιακό δίκαιο, ε, το παραδοσιακό μοντέλο ρυθμίσεων και κανόνων τίθεται να αμφιβόλο. Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι να δώσουμε οριστικές απαντήσεις ε, για να ανοίξουμε το δρόμο για το μέλλον. Θυμάμαι στην προηγούμενη ε, κοινοβουλευτική θητεία ήμουν επικεφαλής μαζί με διάφορους συναδέλφους να ήμουν ας πούμε επιφορτισμένος με το να προβληματιστούμε για την ψηφιακή επανάσταση της κοινωνίας. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε δεν υπήρχε το υπολογιστικό νέφος. Μέσα σε δύο-τρία χρόνια το, τον καιρό δηλαδή που δουλεύαμε εμφανίστηκε το νέφος αυτός. αυτό. Πήραμε λοιπόν αποφάσεις ε, όπου λόγω των κανόνων ε, εμποδίζαμε τον έφος να, να εμφανιστεί. Είχαμε λάθος, έτσι. Προσοχή, προσοχή λοιπόν. Ε, στο να πάρουμε οριστικές αποφάσεις οι οποίες ε, θα μπερδέψουν τα πράγματα για το μέλλον. Επίσης, προσοχή, να μην μπούμε πράγματα εξής αφήξης. Ειδικά στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς πρέπει να, να σταματήσουμε να υπάρχουν εμπόδια και νομοθετική κατακαιρμάτιση. Ε, από ότι, επίσης, έχουμε κατακαιρματισμό μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών, δηλαδή διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες, θα πρέπει ουσιαστικά να διευκολύνουμε την εμφάνιση Ευρωπαίων ε, πρωταθλητών και θα πρέπει να σταματήσει μια δεύτερη κατακερ... Ε, ένας δεύτερος κατακαιρματισμός που είναι πολύ εξειδικευμένο ανάμεσα στον επιγραμμικό κόσμο και στον υπόλοιπο. Ε, οι επιχειρήσεις πουλάνε και στο ίντερνετ και εκτό. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλε αντιφάσει ανάμεσα στου δύο κόσμου. Αυτά. Ε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Λοιπόν, τα θέτω. Θα πρέπει οι δύο επιτροπέ να συνεργαστούν και να αποπειραθούν να βρουν να... Ε, λύσεις. Ε, χαίρομαι εκ των προτέρων για τη συνεργασία με του και όλου και χαίρομαι εκ των προτέρων για αυτή την ευκαιρία που μα δίδεται να διατρανώσουμε την ανάγκη ενό θετικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσει ε, τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Very much, uh, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση να είναι και οι δύο επιτροπέ υπεύθυνε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Περνάμε τώρα στους ισχυτέ. Μέρου Μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, δύο συνάδελφοι. Βλάνκο Λόπε και Γκουγιέρες Πέτο. Όπω θέλετε, με όποια σειρά θέλετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή αυτή, Ήτρε, μιλούσαμε για τη συνεργατική οικονομία. Σήμερα μιλάμε για τις πλατφόρμες. Νομίζω ειλικρινά ότι θα έπρεπε να έχει συνταχθεί μια κοινή έκθεση για τα δύο θέματα. Γιατί κατά την άποψή μου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τώρα, ψηφιακές πλατφόρμες είναι κάτι το οποίο ε, πραγματικά φέρνει επανάσταση στη ζωή μας, όχι μόνο στο ψηφιακό αλλά και στο φυσικό επίπεδο. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ε, χάνει το τρένο. Το λέει και το έγγραφο που συναντεύει την ανακοίνωση. Αναπτύσσουμε εφαρμογέ. Σε αυτό καλοί είμαστε, αλλά σε ό,τι αφορά τι Είμαστε στην τρίτη θέση. ανακαλύπτουμε νέες τεχνολογίες και κόνσεπτ, όμως ό,τι αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των ιδεών, υπολοιπόμεθα των άλλων. 176 πλατφόρμες έχουν μελετηθεί, 25 μόνο από αυτές ήταν ευρωπαϊκές ε, και το 4% ήταν ε, ότι ε, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει κατά την άποψή μου επίση να λάβουμε υπόψη τα πολλαπλά άλλα προβλήματα. Το είχα ξαναπεί ε, όταν συζητούσαμε τη συνεργατική οικονομία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να επανακαθορίσουμε την εργασιακή αγορά για να μην είναι επισφαλής. Υπάρχει ένα θέμα κλειδί που πρέπει να μας απασχολήσει, η φορητότητα της ψηφικής ταυτότητας βέβαια. Υπάρχουν και άλλα θέματα Δηλαδή, πώς θα πετύχουμε τη μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τι μεγάλες Η χρήση των πληροφοριών που συμπηλούν ε, για τους χρήστες τους, οι σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και προμηθευτών, αποφυγή ε, πιθανώς μονοπωλίων, ε, περιστολή κυκλοφορίας ε, μη ενδεδειγμένου παράνομου περιεχομένου και αποβολή καταχρήσεων από τους ε, χρήστες. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον περιμένω τις ε, προτάσεις των εισηγητών. Και επίσης ε, νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητές συνάδελφες, εσείς κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, εμείς ως κοιόδης εισηγητές και εκπρόσωποι των σοσιαλιστών, το πρώτο μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι θέλουμε κανόνες. Όντως έχει γίνει συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μιλάει για καλές πρακτικές και αυτορύθμιση της νέας αγοράς, η οποία αναδύεται. Ε, και όταν βλέπουμε τα ποσοστά τα οποία αυξάνονται στο, σε άλλες οικονομικές περιοχές του πλανήτη, βλέπουμε ότι μας τρώνε όλο και περισσότερο έδαφος και τρώει ε, η ψηφιακή οικονομία όλο και περισσότερο έδαφος από την ε, παραδοσιακή οικονομία. Επομένως, θα πρέπει ε, να ρυθμίσουμε δεν τα πράγματα, να υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τώρα η λεγόμενη αυτορύθμιση αυτής της αγοράς ε, οδηγεί στην εξή κατάσταση. Ε, το να έχουμε διαφορετικές, διαφορετικούς κανόνες, αθέμητο ανταγωνισμό, ε, αθέμητο ανταγωνισμό για τι παραδοσιακέ επιχειρήσει και νέε καταχρήσει. Πρέπει να ρυθμίσουμε, να έχουμε καλούς κανόνε, καλ... ε, ούτως ώστε οι ίδιοι οικονομικοί κανόνε που δραστηριοποιούν στον ίδιο χώρο να διέπονται από του ίδιου κανόνε και να δώσουμε ε, καλές ευκαιρίες στους εργαζόμενους και οικονομική ανάπτυξη. Όντω, ε, ορισμένοι λένε, και εγώ πιστεύω σε αυτό, ότι η συνεργατική οικονομία, η νέα ψηφιακή οικονομία μπορεί να εκδημοκρατικο κοπήσει την ε, γενική οικονομία. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχουν δίκαιοι κανόνες, ξεκάθαροι κανόνες. Το ξέρουμε όλοι μας. Και στοιχηματίζουμε ε, σε μια φιλόδοξη πρόταση που θα πρέπει να προτείνει η, κοινοτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προτείνει και μια καλή νομοθεσία. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε. Σωστό είναι αυτό. Αλλά έχουμε αρκετή εμπειρία τώρα. Προφανώς και άλλες περιοχές οικονομικές του πλανήτη έχουν τέτοια εμπειρία, αλλά κυρίως η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και κυρίως η Ευρωζώνη έχει εμπειρία για να φτιάξει βασικούς κανόνες. Σωστό είναι ότι η νέα οικονομία μπορεί να, δώσει, να οδηγήσει σε νέες καταχρήσει. Επομένως, η υποχρέωσή μας είναι να προλάβουμε, να μην υπάρξουν αυτέ οι καταχρήσεις, ε, να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, να προστατεύσουμε τον ε, εργαζόμενο και επίσης θα πρέπει να υπάρχει η έννοια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης ε, για τις εταιρείε οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτές τι ψηφιακέ πλατφόρμες. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να ρυθμίσουμε την ε, προστασία, να υπάρχουν κανόνε δηλαδή στην προστασία του καταναλωτή. Σε μια οικονομία, σε μια ενιαία αγορά, όπου και η παραδοσιακή οικονομία έχει βάζει πολλές ε, προκλήσεις για να προστατεύσουμε τον ε, καταναλωτή. Φανταστείτε, πολλό δε μάλλον στην ψηφιακή οικονομία. Πόσες περισσότερες προκλήσεις ε, υπάρχουν. Ε, με βάση τους παραδοσιακού κανόνες που έχουμε για την προστασία του καταναλωτή, ε, σε ένα κόσμο γεμάτο από διαμεσολαβήσεις και διάμεσους κτλ, θα πρέπει οι καταναλωτές να ξέρουν τι τους, περι... τι τους ξημερώνει, τι κανόνες υπάρχουν. Θα πρέπει να ξέρουμε τη διαφορά ανάμεσα στον αυτοαπασχολούμενο και στον εργαζόμενο, ε, σε αφεντικό, σε... για λογαριασμό κάποιου άλλου στις ε, ψηφιακές ε, πλατφόρμες. Ε, ίδιοι κανόνες, λοιπόν, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις νέες προκλήσεις, όπως λέει ο συνάδελφος από την Ήτρε. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, τελειώνω. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το rating ε, για την ε, αξιολόγηση δηλαδή, των χρηστών ε, από τους χρήστες ε, των πλατφορμών αυτών. Γιατί υπάρχει μια φαιά ζώνη, ας πούμε, και εκεί ακριβώς δημιουργούνται νέες, νέες απάτες. Ο προηγούμενος συναδελφός μίλησε ένα λεπτό λιγότερο, αλλά δεν μπορούν οι σχεδόν να μιλάνε πάνω από τρία λεφτά. Όχι, όχι, θα σταματήσω εδώ, εντάξει. Περνάμε τώρα στην ECR. Βαν Βόσιους, Κάθεσαι σε ένα μέρος ε, κάπως απίθανο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πράγματι, κάθομαι σε λάθος θέση, λέει η κυρία Φαν Μπόσεντ. Είμαι μέλος της Επιτροπής Ήτρε αλλά και της Επιτροπής ΙΜΚΟ ε, και βρίσκομαι εδώ ο κοιόδηση εισηγήτρια για την ECR εκ μέρου τη ΣΥΤΡΕ, όμω όπω σα είπα συμμετέχω και στην ΙΜΚΟ. Και ελπίζω ότι και από τις δύο, από τις δύο γωνίες θα μπορέσω να εξετάσω το έγγραφο που θα προκύψει. Πιστεύω ότι με το γενικό αυτό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προσπάθησε να σφιγμομετρήσει από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δει κατά πόσο υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης ε, σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο ένωσης ε, για κάποιες πτυχές του, του θέματος αυτού. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες δεν μπορούν ε, να μπουν όλες στο ίδιο σακί. Κάποιες δραστηριότητες μπορούν να θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία Spotify, Amazon, ε, Airbnb. Δεν λέω ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά ίδιοι οι κανόνες. Κάποια από τα ζητήματα των επιγραμμικών πλατφορμών έχουν ε, ήδη καλυφθεί, για παράδειγμα, από την οδηγία για τα οπτικοδοστικά, για τα δικαιώματα του δημιουργού, ε, το πακέτο των τηλεπικοινωνιών κλπ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν θα σας κάνει εντύπωση αυτό που θα πω, να μην παρεμποδίσουμε μέσω καινούριων κανόνων την καινοτομία ή την εμφάνιση άλλων παικτών. Πρέπει οπωσδήποτε να ενθαρρύνουμε ε, την, το επιχειρήν, όπως κάνουμε και στους ε, πιο κλασικούς τομείς. Πολλές πλατφόρμες που γνωρίζουμε σήμερα είναι πλατφόρμες που προέρχονται από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, έχουμε λοιπόν ως Ευρώπη μια τρομερή καθυστέρηση στους τομείς αυτούς και πρέπει οπωσδήποτε να καλύψουμε την καθυστέρηση αυτή. Πολλές φορές ε, θέλουμε να ρυθμίσουμε σε υπερβολικό βαθμό και αυτό μερικές φορές γυρίζει εναντίον μας και πρέπει να το αποφύγουμε. Σε κάθε περίπτωση και δεν χρειάζεται να κάνουμε αντιγραφή και επικόλυση ε, των δραστηριοτήτων. Ε, αν για παράδειγμα κάποιος μέσω Airbnb κάνει κράτηση για ένα δωμάτιο, δεν πρέπει να τοποθετείται στη ίδια κατηγορία με τον ιδιοκτήτη ενός ε, ξενοδόχου που έχει 120 δωμάτια να διαθέσει. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι πλατφόρμες αυτές να έχουν και εκείνες τις ευθύνες τους ως Προ την προστασία του καταναλωτή, να μην χάνεται αυτή η ευθύνη. Όσον αφορά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε σήμερα, νομίζω ότι ήδη ε, διαφαίνεται καθαρότατα ότι είναι μια καλή ισορροπία, είναι, θα είναι μια ωραία περιπέτεια και με πολύ χαρά την ε, περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τηρήσατε και το χρόνο σας. Εκ μέρους των, ε, των φιλελευθέρων έχω τον Κόραν Φανιούενχόζεν. Θα μιλήσει εκ μέρους των δύο σκιωδών. κυρία, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Και η κυρία Καλής και η κυρία Ελίνα δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα στη συνεδρίαση αυτή, οπότε θα τα προσωπήσω και τις δύο. Καταρχάς, η εκθέση αυτή για τις επιγραμμικές πλατφόρμες έρχεται σε μια χρονική στιγμή που γίνονται συζητήσεις για διάφορα τομεακά νομοθετήματα, EVMS, ε, μεταρρύθμιση πνευματικών δικαιωμάτων, ε, τηλεπικοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό για την Άλντε να δώσουμε τη δουλειά μας περισσότερο καθοδήγηση και όχι ε, αμφιλεγόμενα νομοθετήματα και αντιπαρατηθέμενα το ένα προς το άλλο. Ένα σημαίνει σαφές, ε, το πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν θα πρέπει να υπονομευθεί και ιδίως το άρθρο 14 για την περιορισμένη ευθύνη των διαμεσολαβητών, το διαδικτύο και το άρθρο 15 για, τη, για μη γενική υποχρέωση παρακολούθηση. Υπάρχουν τα ζητήματα επίση του κατακαιρματισμού για τον τρόπο με τον οποίο η οδηγία θα εφαρμόζεται σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι καλή η ευκαιρία εκθέση αυτή, γιατί θα παράσχει καθοδήγηση ακριβώ από αυτή τη εφαρμογή, τη υλοποίηση. Η Κομισιόν επίση δεσμεύτηκε στο δεύτερο ήμιση του 2016 να διαρευνήσει την ανάγκη καθοδήγησης για την ευθύνη των πλατφόρμων όταν υιοθετούν ε, εθελοντικά μέτρα για την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου. Ενδιαφέρον θα ήταν να ακούσουμε ε, μια επικαιροποιημένη τοποθέτηση της Κομισιόν επ' αυτού. Ένα άλλο σημείο αφορά τη διαφάνεια και την δικαιοσύνη. Σημείο δράση για την Κομισιόν στην νομοθετική πρόταση για την προστασία των καταναλωτών και τη σχετική συνεργασία είναι η βελτίωση τη διαφάνεια. Όμω, στην πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει νέες εξουσίες στις αρχές αυθαίρετα να μπορούν να κλείνουν ε, ιστοσελίδες ε, ε, ή, να, ή τομείς, ονομασίες τομείς. Αλλά αυτά δεν είναι καλά. Ούτε για τη διαφάνεια, ούτε για την καινοτομία. Άρα, έχουμε κάποιες ανησυχίες σχετικά. Και που πιστεύουμε ότι χρειάζεται τη διαφάνεια πάντως, είναι στα business to business στο επιγραμμικό περιεχόμενο. Πολλέ φορέ οι μικρέ επιχειρήσει ε, βασίζονται στι πλατφόρμες για τι επιχειρηματικέ του δραστηριότητε. Θα πρέπει να υπάρχουν ό,τι και προποθέσει, ιδίω σε ό,τι αφορά αναβαθμίσει ε, και επικαιροποιήσει. Αυτό θα πρέπει να είναι διαφανή για να γνωρίζουν οι επιχειρήσει τι να περιμένουν όταν βασίζονται σε πλατφόρμες. Σας ευχαριστώ ε, και προσβλέπω να συνεργαστώ, μάλλον προσβλέπουν και οι δύο συνεισηγήτριες, τις οποίες εκπροσώπησα, να συνεργαστούν με τους δύο συγητές. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε κόρα. Όπως βλέπω τώρα στον κατάλογό μου, ο τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί ένα πολύ σημαντικό ερώτημα για αυτή την έκθεση. Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες που έχουν τώρα δύναμη και προσφέρουν υπηρεσίες. Που δεν μπορούμε ε, να πούμε ότι οδηγούν ε, στη βελτίωση αγοράς με το Facebook, το Google, την Apple, που έχουν πολύ μεγάλη δύναμη ε, στην αγορά. Και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και σε ό,τι αφορά την πολιτική και τη δημοκρατία. Και δεν το βλέπουμε ίσως τόσο έντονα σε άλλους τομείς. Άρα θα πρέπει ακριβώς ε, αυτό να βοηθήσουμε με αυτή την ε, νομοθεσία, να δώσουμε δηλαδή δυνατότητες βελτίωσης σε αυτές τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Όχι όμως ε, να αφήσουμε αυτή τη δύναμη σε αυτές τις λίγες πλατφόρμες, γιατί αν αφήσουμε τα πράγματα έτσι τις επόμενες δεκαετίες... δεν θα κάνουμε κανένα χατήρι, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε ε, να προωθήσουμε, να βελτιώσουμε τη θέση μας. Ε, θα πρέπει η ευρωπαϊκή βιομηχανία όμως να ειδωθεί και από κοινού και με τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Από πολιτικής, δημοκρατικής πλευράς είναι πολύ επικίνδυνο λίγες επιχειρήσεις, μόνο λίγες επιχειρήσεις, να έχουν τόσο μεγάλη επιρροή και να μπορούν να επηρεάζουν τις πολιτικές διαδικασίες και την κοινή γνώμη, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και ε, κατά το παρελθόν είδαμε με την επανάσταση των ε, ε τηλεπικοινωνιών να, προστατεύσουμε με διάφορες διατάξεις ε, και την κοινή γνώμη. Θα πρέπει από πολιτικής πλευράς λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση να προβληματιστούμε και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με αυτές τις πλατφόρμες. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ αποφασιστικά βήματα και όχι κάτι λίγο θα πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ καλά. Όχι μόνο τα, ε, μάλλον τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών βιομηχανών και επιχείρησεων, αλλά και των ευρωπαίων πολιτών, που κατά την άποψή μου συμβαδίζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν είχα στον κατάλογο μου και συγγνώμη την κυρία Τζούλια Ρέντα, τους πράσινους της ΣΥΜΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Ράιμοντ είπε διάφορα πράγματα για τη σημασία των ε, βασικών θεμάτων του δίκαιου ανταγωνισμού και της ε, διαφάνειας. Είμαστε σε ειδική κατάσταση, γιατί πολλές από τις νομοθετικές προτάσεις της, ε, της Κομισιόν στην ανακοίνωση για τις πλατφόρμες έχουν ήδη παρουσιαστεί και εμείς συνεργαζόμαστε σε διάφορες επιτροπές από αυτών για τον κώδικα, για την ε, IDMS, ε, για την ε, ιδιωτικότητα, προστασία των καταναλωτών. Δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε λοιπόν τις προσπάθειες που γίνονται αλλού. Αν θέλουμε να γεννήσουμε προστιθέμενη αξία με αυτή την πρόταση, να εστιάσουμε σε κάποιες από τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν σε αυτή την ανακοίνωση και που εκκρεμούν ακόμα. Η Κομισιόν μιλάει για τη δημιουργία ενιαίων διαδικασιών, ε, για να κλείνουμε πλατφόρμες, για την ε, περιορισμένη ευθύνη, για τη διαλειτουργικότητα, ε, για τη διαφάνεια, σχέσεις B2B και για την χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από την αναζήτηση σε μηχανή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια κοινή θέση για τις πλατφόρμες στην έκθεση για την ψηφιακή κοινή αγορά και αυτά όλα θα πρέπει να τα έχουμε ως αφετηρία. Έχουμε ήδη διατρανώσει κάποιες βασικέ θέσει και απόψει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε δηλαδή στην εφαρμογή και των, της νομοθεσία, κυρίω ε, στο δίκαιο του καταναλωτή, όπου πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, να υπάρχει αποτελεσματικό ανταγωνισμό μεταξύ των πλατφορμών, ε, από διαφορετικού τομεί, να μην έχουν αλυσιδωτέ επιπτώσει στου καταναλωτέ, να μπορούν να αλλάζουν από πλατφόρμα σε ε, πλατφόρμα, να μην υπάρχουν στρεβλώσει τη αγορά ε, μέσω των υποχρεώσεων ε, για επιχορήγηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών μοντέλων και τέλος ε, η περιορισμένη ευθύνη της οδηγίας. Η Κομισιόν είπε στην ανακοίνωσή της, δεν θέλω να αγγίξω αυτό το τελευταίο, θέλω να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι αυτή η αρχή για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την, το να είναι ανοιχτό το, το ίντερνετ, για την νομική ασφάλεια και για την κοινοτομία. Αν θέλουμε περισσότερες ευρωπαϊκές πλατφόρμες σε αυτόν τον τομέα που να είναι επιτυχής σε παγκόσμια κλίμακα και παράλληλα να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, τότε οι αρχές της οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η βάση και πρέπει να τις διατρανώσουμε και να τους προστατεύσουμε. Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τους βασικούς εισηγητές, όλα όσα είπατε. Ο Ντάνιελ Ντάλτον από την ECR για την ΙΜΚΟ στέλνει ένα σύντομο σημείωμα στους συναδέλφους του και το έχει δώσει μάλλον στην κυρία Αντλίν Βαν Μπόσεν. Διαβάστε το σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ, οπότε εγώ θα διαβάσω την ε, δήλωσή του. Είναι πάρα πολύ σύντομη. Αυτό λοιπόν που θα ήθελε να πει προς τους εισηγητές αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήταν ευπρόσδεκτη και ε, την περιμένουμε πολύ καιρό. Ήταν σωστή στην αξιολόγησή της ότι πρέπει ότι η η υπερβολική ρύθμιση δεν είναι καλή. Πρέπει να σκεφτούμε ε, πολύ καλά πριν ε, αφήσουμε κατά μέρο παλιά νομοθεσία και εισάγουμε νέους κανόνες. Ε, δεν ε, πρέπει να καταστρέψουμε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην, και διαδικτυακών τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ενώση πρέπει να υπάρχουν συγκρίσιμοι κανόνε ε, για συγκρίσιμε υπηρεσίε, όμω αυτό έχει ερμηνευτεί με διαφορετικού τρόπου από τα κράτη-μέλη και θα ήθελε να ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί αυτού τι έχει σκοπό να κάνει. Ε, το Airbnb θεωρείται το ίδιο πράγμα με ένα κλασικό ξενοδοχείο, για παράδειγμα. Πρέπει να έχουμε μια καινοτόμο προσέγγιση σε μια τόσο μεταλα... Ε, τεχνολογία. Μπορεί ε, να δημιουργήσουμε μια μαύρη ψηφιακή οικονομία αν ε, δεν κάνουμε τη διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιγραμμικών πλατφορμών γιατί έχουν εντελώς διαφορετικές μορφές και μεγέθη. Ε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα μικρή κοινότητα ε, επιχειρήσεων ε, που θα δράμε το δικό της τρόπο. Υπάρχει η οδηγία EVMS ε, για την οποία κάποιοι θεωρούν ότι δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση στις πλατφόρμες και από άλλους θεωρείται μια καλύτερη και πιο ρεαλιστική προσέγγιση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είναι όμως ε, μια πολύ μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις πλατφόρμες αυτές και αναμένει εναγωνίως τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω την Προεδρία τώρα στην κυρία Φόρντ. Λοιπόν. Sean Kelly, Nicola Dante, Pascal Arimont, Sabine Verheyen, um, Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο και η κυρία Γκέπχαρτ, εκτός από όλους όσους ανέφερα που θα πάρουν το λόγο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μισελ Μπόνι. Ευχαριστώ πολύ. Τρία σημεία. Καταρχάς, η ευθύνη των διαμεσολαβητών. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να το συζητήσουμε και να έχουμε και αυτορυθμιστικά μέτρα για να αποφύγουμε τις αθέμητες πρακτικές, ε, το παράνομο μη ενδεδειγμένο περιεχόμενο. Καλή η νομοθεσία, σημαντικό όμω είναι ταυτόχρονα να αποφευθεί και ο κατακαιρματισμό στην Ευρώπη. Και πρέπει να είναι αυστηροί οι κανόνες για την αυτορύθμιση και την ρύθμιση εν γέννη στην Ένωση. Δεύτερον, θα πρέπει, πιστεύω, να δούμε ότι υπάρχουν ε, αρκετοί διαφορετικοί τύποι πλατφορμών και πρέπει να το λάβουμε υπόψη κατά την εκπόνηση της ε, Υπάρχουν τηλεϊατρικές πλατφόρμες ε, που έχουν να κάνουν με την υγεία ε, ή άλλε που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα για μας που είμαστε χρήστες των πλατφόρμων και τι μελλοντικέ εξελίξεις στην παροχή των λόγων υπηρεσιών. Και το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφόρμων. Κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είμαι βέβαιος για το κατά πόσο γι' αυτό θα παιδηθούν διαφορετικοί κανόνες. Αλλά αν συζητάμε για όλα αυτά τα είδη πλατφορμών θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και δεν μπορούμε να έχουμε μια νέα προσέγγιση για όλες τις πλατφόρμες. One size fits all. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σον Κέλλη τώρα. Ευχαριστώ συγχαρητήρια και στους δύο για την επανεκλογή σας. Μιλήσαμε, μίλησαν άλλοι συνάδελφοι, για τα τεράστια πλεονεκτήματα, τις τεράστιες ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Και κάποιος άλλος είπε ότι ε, το μερίδιο της ε, ευρωπαϊκής, το μερίδιο της αγοράς από πλευράς Ευρώπης είναι 4%. Αυτό είναι ένα κατηγορό για την Ευρώπη. Και όσοι αγαπούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να την προωθήσουμε, εάν δεν αλλάξουμε ε, αυτό το ποσοστό δεν μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε και ότι είναι επιτυχημένοι. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητέ σε ορισμένου τομεί, στου στόχου για την κλιματική αλλαγή, Φερρυπίν, για τη μείωση των εκπομπών κτλ. κτλ. Θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχο στόχο και εδώ. Να έχουμε 30% τη αγορά μέχρι το 2030 και να εξασφαλίσουμε ότι δεν βάζουμε εμπόδια ε, στο δρόμο των πλατφορμών όπως κάνανε και οι προηγούμενοι ομιλητές. Αν τα καταφέρουμε, αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, θα τα καταφέρουμε, θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Ε, Τάντι. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις. Εγώ ως εισηγητής για τη συνεργατική οικονομία είχα τη δυνατότητα αυτή την περίοδο να αναλύσω κάποιες πτυχές που αφορούν τις πλατφόρμες. Και μία πτυχή αφορά την ε, συνεργατική οικονομία, αλλά και πολύ περισσότερο, πολύ πέρα από, αυτά, από αυτήν. Υπάρχουν διάφορα προβληματικά σημεία που θα πρέπει να αναλύσουμε εμεί αυτό το γενικό θέμα των πλατφορμών. Τα απαριθμώ γρήγορα. Καταρχά το θέμα του ανταγωνισμού και τη ε, τάση τη μονοπωλιακή που βλέπουμε στι πλατφόρμε. Τάση να δημιουργούνται μονοπόλια. Όπω όλε τι αγορέ υπάρχει αυτή η τάση, α πούμε, αν δεν υπάρχουν ρυθμίσει και κανόνε. Και στο σύστημα λοιπόν των πλατφορμών αρχίζει να διαφαίνεται μία μονοπωλιακή τάση. Σκέφτεται κάποιε μεγάλε πλατφόρμε, α πούμε, που είναι εντελώ μονοπωλιακέ αυτή τη στιγμή στον κόσμο, όχι στη χώρα του, στον κόσμο σε κάποιου τομεί, α πούμε, τη οικονομία μα. Επομένω, το θέμα του πώ θα καταφέρουμε να αποφύγουμε στο σύστημα της ψυχιακή οικονομία ε, και στι πλατφόρμες να δημιουργηθούν μονοπόλια και κλείσιμο τη αγορά. Πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αγορά να μπουν και άλλε περισσότερε επιχειρήσει. Δεύτερο θέμα. Το θέμα τη φήμη που έχει κανεί online. Ε, μετράει πάρα πολύ και για τον πάροχο υπηρεσιών και για του πελάτε. Η φήμη είναι μια τεράστια αξία, μια... ένα τεράστιο θέμα. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ξεκάθαρου κανόνε στην αγορά. Για το πώ χτίζεται μια φήμη, α πούμε, με ποιου αλγόριθμου, α πούμε, γίνεται Και αυτό το στοιχείο, ας πούμε, ανήκει σε κάποιον, μπορεί να το μεταφέρει, ας πούμε, ε, είναι ε, στην κατοχή, ας πούμε, της πλατφόρμας ή του πελάτη, ας πούμε. Είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο θα πρέπει εμείς να αξιολογήσουμε. Στις ΗΠΑ ε, προκύπτει ξεκάθαρα η εξιστάση. Αρχίζουν να αναλύουν και να βλέπουν φαινόμενα διακρίσεων στο εσωτερικό των πλατφορμών. Παραδείγματο χάρη, ε, αναφέρονται πράγματα, ας πούμε, για το χρώμα του, α, του, του, του καθενό Προσοχή, προσοχή, όχι τέτοιε αναφορέ. Έχει να κάνει με την ελευθερία μα. Επίση, διαχείριση των πλατφορμών. Ξέρουν τα πάντα. Τι φιλοδοξίε μα, τι τάσει μα, τι, θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Ε, το φίλο μα. Ε, Προφανώ πρέπει να έχουν κανόνε, ε, ούτω ώστε οι πλατφόρμε να μην κάνουν ό,τι θέλουν. Να εξασφαλίζονται οι καταναλωτές. Ε, γιατί μιλάμε για δεδομένα που αφορούν τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις ε, αυτές για τους εισηγητές και για όλους μας. Ε, ώστε να δημιουργήσουμε ευνοϊκές προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί αυτός σημαντικός τομέας της μελλοντική οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ, Βίκη είμαι εισηγητής για μια έκθεση που αφορά και τα προϊόντα και τις εξαποστάσεις πωλήσει και θα ήθελα και εδώ να πω ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε κριτήρια. Συμφωνώ με κάποιους συναδέλφους που λένε ότι αν βλέπουμε ήδη σε αυτό το τομέα μονοπωλιακές καταστάσεις πώς αυτές τις ε, ε, μονοπωλιακές ε, συνθήκες ή με αυτές τις επιχειρήσεις και την παροχή πρέπει θα τις αφήσουμε σε χέρια Αμερικανών ή τέλο πάντων τρίτων. Βέβαια, μονοπόλιο είναι μονοπόλιο μέχρι να βρεθεί κάποιος να κάνει καλύτερα τα πράγματα. Η νοκια είναι ένα καλό παράδειγμα για το τι, τι μπορεί να συμβεί και στις συζητήσεις ε, που άκουσα ε, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες βασικές γραμμές γύρω από τις οποίες πρέπει να κινηθούμε για τις ε, πλατφόρμες. Πλατφόρμες είναι ένα ένα εργαλείο και για την έκθεση τη δική μου, δηλαδή για τις εξαποστάσεις αγορές προϊόντων. Σίγουρα προσφέρουν πάρα πολλά, το γνωρίζουμε όλοι. Το θέμα είναι ανεξαρτήτως του τομέα που θέλουμε να ρυθμίσουμε, αν εκπονούμε κανόνε, οι κανόνε αυτοί πρέπει να είναι απλοί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδίω στην ψηφιακή αγορά. Ευνόητοι, ε, απλοί κανόνε για να υπάρχει ανταγωνισμό. και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν είναι εναρμονισμένοι αυτοί οι κανόνε. δηλαδή να έχουμε νέου κανόνε για τα 28 κράτη-μέλη. Αν αυτό δεν το πετύχουμε, να έχουμε νέου κανόνε δηλαδή για τα 28 κράτη-μέλη, ποιον βοηθούμε τελικά, βοηθούμε μόνο αυτού που θέλουν πιο ισχυρά μονοπόλια ακόμα με τις διαφορετικούς ε, ε, κανόνες και ρυθμίσεις, ποιος μπορεί να ε, τα φέρει πέρα καλύτερα. Οι μονοπρόσωπες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις ή οι μεγάλοι όμιλοι. Οι μεγάλοι όμιλοι ε, βλέπω και την κυρία Γκέπχαρτ που φαντάζομαι θέλει να πει κάτι επ' αυτού. Ε, δεν πολύ συμφωνούμε κάποιε φορέ, αλλά τέλο πάντων. Τι θα κάνουμε την ε, προστασία των καταναλωτών. Μπορεί να είναι ένα επιχείρημα η προστασία των καταναλωτών, ε, γιατί θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Το θέμα είναι αυτά τα δικαιώματα για την προστασία των καταναλωτών, πόσο υψηλή θέση πρέπει να έχουν, το θέμα είναι να είναι ενημερωμένοι οι καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και αυτά τα δικαιώματα να ισχύουν και να προστατεύονται. Ευχαριστώ. Η Σαμπίν Φερχάιν, ευχαριστώ για τις μονοπωλιακές δομές, ε, την προστασία των καταναλωτών, ε, υπόθηκαν πολλά ήδη. Για τον τομέα επίσης και της ευθύνης ε, υπόθηκαν αρκετά σε ό,τι αφορά την ε, ρύθμιση για τις πλατφόρμες, το liability, για τους ενδιάμεσους, όλα αυτά η ευθύνη είναι σημαντικό. Ε, νομίζω ότι έχουμε σωστές διατάξεις στην οδηγία. Βέβαια θα πρέπει να ορίσουμε ξεκάθαρα το πού ξεκινάει η ευθύνη. Εγώ προσωπικά ε, μια ενεργή πλατφόρμα που η οποία πραγματικά παρέχει, διαθέτει προϊόντα, πώς διαχωρίζεται από έναν ενδιάμεσο. Και σίγουρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι από ποια ε, από ποιο είμαι και μετά είμαι ένας ενεργός παίκτη ε, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ε, διαθέτω. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσα να αναφέρω. Αν, ας πούμε, ε, κάποιος κάνει διαφημίσεις συγκεκριμένα ε, στην πλατφόρμα για συγκεκριμένα. Ε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το περιεχόμενο, αν είναι παράνομες, ή παράνομο ή νόμο το περιεχόμενο. δεν μπορεί μια πλατφόρμα να ισχύσει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Πρέπει να βρούμε κατάλληλες ρυθμίσεις πιο καλά προσαρμοσμένες. Γκέπχαρτ. Η Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους δύο για την πολύ καλή τους ε, δουλειά. Με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια και συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να παραμείνουμε συνεκτικοί και συνεπείς στην πολιτική μας. Το να είσαι κανείς συνεπής στην πολιτική σημαίνει ότι η συνεργατική οικονομία και οι πλατφόρμες δεν θα πρέπει να ειδωθούν ξεχωριστά μεταξύ τους για τη διαφοροποίηση μεταξύ του τι είναι πλατφόρμα και του τι είναι sharing economy, συνεργατική οικονομία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολο να κάνουμε τη διάκριση. Θα πρέπει λοιπόν να ε, φροντίσουμε να αποφύγουμε ασυνέπειες κ. Σαριμών πολύ καλά τα είπε, ότι πράγματι δεν συμφωνούμε και πολύ συχνά στην Επιτροπή μας, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας εδώ, ότι φυσικά είναι το καλύτερο να έχουμε κοινή νομοθεσία, κοινού κανόνες και δεν θα πρέπει οι κανόνες που ήδη ισχύουν στα κράτη-μέλη να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Και εκεί νομίζω ότι έγκυται τη διαφωνία μας, γιατί εσεί λέτε ότι ναι, ε, αν ε, κάνουν λιγότερα κάποια κράτη-μέλη, αλλά μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, ίσως πρέπει να μην. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί οι καταναλωτές ε, έχουν να κάνουν... Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα θέματα τη παράδοση. και πρέπει να δούμε τι παράδοση ισχύει ε, για τους καταναλωτές τι ήθη και έθιμα έχουν. Και σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες, και αυτό πρέπει να ισχύσει, γιατί θα εμπιστευτούμε τις πλατφόρμες περισσότερο μόνο αν φροντίσουμε να νιώθουν καλά οι καταναλωτές, ε, πολύ καλά, να νιώθουν άνετα με τις πλατφόρμες, αν φοβούνται, αν φοβούνται ότι τα δικαιώματά τους θα περιοριστούν. Δεν θα τις χρησιμοποιήσουν αυτές τις πλατφόρμες. Και νομίζω ότι αυτό πάντα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επιμείνω στο τεράστιο δυναμικό που ε, σημαίνει η οικονομία των πλατφορμών ε, και ότι υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρξει ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον που θα δώσει τη δυνατότητα της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων και των ε, ευρωπαϊκών πρωταθλητών. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να βασιστούμε, να δουλέψουμε ιδίω στην εμπιστοσύνη και την ομιμότητα γιατί ε, πάρα πολύ είναι μικρό το ποσοστό, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που έχει εμπιστοσύνη στα κοινωνικά δίκτυα και πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη είναι το, κλει, το, το κλειδί για την επιτυχία των, ε, ψηφιακών υπηρεσιών. Θα μπορούσε βέβαια περάσει μέσα από διάφορα στοιχεία τα οποία πρέπει να δουλέψουμε, όπως για παράδειγμα υποχρέωση ενημέρωσης ε, σαφούς ε, των ε, καταναλωτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω αυτών των πλατφορμών, ώστε να υπάρχει ασφάλεια Επίσης πρέπει να ασχοληθούμε με τους μηχανισμούς πιστοποίησης, ε, σχολείων ε, και απόψεων, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της φήμης ε, στο διαδίκτυο, να υπάρξει μια συνεργασία εκ των προτέρων των πλατφορμών με τις διοικήσεις. Τώρα, με την ιδιότητά μου ως εισηγήτρια σκιώδη της Επιτροπής Απασχόλησης, θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι αν θέλουμε να, να επιτρέψουμε την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας ε, γενικότερα, πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ως προς τις αρμοδιότητες για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στους πολίτες, στους εργαζόμενούς μας ε, να ε, έχουν την πλέον κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από λίγες μέρες παρευρέθηκα στην, ε, σε μία ομιλία του Ρωμάνου Πρόντι. Ε, επίσης ένας, γινόταν, ένας άνθρωπος γινόταν ακαδημαϊκός και έκανε, έβγαλε μία ομιλία. Μιλούσε για τις οικονομικές δυσκολίες, ε, τη δυσκολία που έχουμε να περάσουμε από την ύφεση στην ανάπτυξη. στι μεγάλε αλλαγέ στην Ευρώπη, ε, πάντα ξεκινούσαν, άνοιγαν νέε εποχέ, νέε οδοί. Ξε, ε, μην ξεχνάτε, ας πούμε, την, α, τις ανακαλύψεις, ας πούμε, στο 15ο αιώνα ή τον τρόμο του μεταξιού, ας πούμε, που οδήγησαν σε μεγάλη ανάπτυξη εν συνεχεία στην Ευρώπη για αιώνες. Όμως, εδώ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Για το ίντερνετ, ο Ρωμάνο Πρόντι είπε ότι αυτό που έγινε είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες και μίλησε για τους ε, κινδύνους που δημιουργούνται από αυτές τις πλατφόρμες ε, γιατί τελικά αναπτύσσονται αλλού και ποτέ δεν είναι πρωταγωνίστρια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, εδώ δεν μιλάμε για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Να το θυμίσω στον προλαλήσαντα αυτό, έτσι. Μιλάμε για θέματα αγοράς, μιλάμε για θέματα εξουσίας την επόμενη ε, Δευτέρα θα, θα γιορτάσουμε την ε, Παγκόσμια ημέρα ε, προστασίας των δεδομένων. Είναι η νέα γεωγραφία της εξουσίας. Το θέμα είναι ποιος αλήθει τα δεδομένα. Αυτός θα έχει την εξουσία. Τις προάλλες, ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ, αυτός που δημιούργησε το Facebook, ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει στις αμερικάνικες ε, εκλογές, δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος σε τέσσερα χρόνια. Ε, μετά από φήμες που κυκλοφορούσαν επί μέρες, ανακοίνωσε ένα νεαρό παιδί, ας πούμε, ε, ότι δεν θα κατέβει στις ε, προεδρικές εκλογές στην Αμερική. Μιλάμε για τέτοια φαινόμενα. Για... Κυκλοφορούσαν φήμες ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Καταλαβαίνετε τι ε, θέματα παίζονται εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για την ελευθερία, ας πούμε, επιλογής των καταναλωτών. Ε, η Αμερική ανακαλύφθηκε όχι από μια νεοφύη επιχείρηση, ας πούμε, με μια βαρκούλα, ας πούμε, αλλά από μια ε, απόφαση κυβερνητική, από τις πιο σημαντικές κυβερνήσεις εκείνης εποχής, να κάνει ε, αυτό το βήμα. Ας διερωτηθούμε λοιπόν, εμείς έχουμε το 4% ας πούμε τον, α, της αγοράς ας πούμε στις πλατφόρμες. Το υπόλοιπο το έχουν άλλοι. Εάν δεν ασχοληθούμε σοβαρά, θα έχουμε απίστευτα βάσανα στο μέλλον. Θα την οπαθήσει η Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δουλειά σας. Ε, στο πλαίσιο της συνεργατικής ε, οικονομίας ε, ασχολούμαστε και εμείς με πολλά σχετικά θέματα στην ΙΜΚΟ και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τα τεράστια ωφέλη που προέρχονται, που υπάρχουν για την κοινωνία, για τους καταναλωτές και τις οικονομίες λόγω των πλατφορμών. Αν θέλουμε ε, οι διαδικτυακοί γίγαντες να ε, αναπτυχθούν στην Ευρώπη πρέπει να μην κόψουμε τα πόδια των ε, ψηφιακών μωρών για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Υπάρχει ήδη αρκετή ρύθμιση με την οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι πλατφόρμες αυτές. Όσον αφορά τώρα την ευθύνη των ενδιαμέσων, υπάρχει ένα ζήτημα με την μουσική και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, αλλά αν προσπαθήσει απλώς να αντιγράψει και να επικολλήσει τους ε, ε, κανόνες σε μια πλατφόρμα, για παράδειγμα, που ε, παρέχει πραγματικό υλικό, όχι ψηφιακό, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν τα μηνύματα μέσω κινητών, υπάρχουν τα, τα μηνύματα μέσω facebook, υπάρχουν 100.000 μηνύματα που μπορούμε να στείλουμε σε σχέση με το τηλεφώνημα που μπορώ εγώ να κάνω στη μαμά μου. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν αυτήν την τεράστια πλειονότητα επιλογών που υπάρχουν. Ναι, θέλω κι εγώ οι ψηφιακέ αγορέ να την κάνουν τη ίδια μεταχείριση με τι άλλε αγορέ, όμω μερικέ φορέ είναι διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με του καταναλωτέ και έχουμε και ένα πραγματικό πρόβλημα με τα δεδομένα ειδικότερα σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος εκεί στο βάθος της αίθουσας. Ε, έχουμε δαπανίσει πάρα πολύ ενέργεια εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο για το GDPR ε, σε ολόκληρη ε, την Ευρώπη. Προσπαθεί ο κόσμος να εφαρμόσει αυτούς τους κανόνες για, τα, για την προστασία δεδομένων, να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε να δουλέψουν και να μην χρειάζεται να τα ξαναγράφουμε από την αρχή σε κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε στο Κοινοβούλιο. Ας αρχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε πλέον κατάλληλη την νομοθεσία που έχουμε προς εφαρμογή και όχι κάθε φορά καινούρια νομοθεσία γιατί αυτό πνίγει την καινοτομία. Γιέζη, σου δίνω το λόγο για να ε, ολοκληρώσεις. Συμφωνώ. Βίκη, απολύτως με τη δήλωσή σου η δική μας ευθύνη ε, ως νομοθέτη είναι πολύ απλή να δημιουργήσουμε το απαραίτητο πλαίσιο, τις απαραίτητες συνθήκες, το απαραίτητο περιβάλλον ε, για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε ε, την ανάπτυξη ε, όλων των επιγραμμικών πλατφορμών στην Ευρώπη. Είναι τεράστια ευθύνη. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Καλό είναι να είμαστε όσο το δυνατόν ταχύτεροι, αλλά μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο ε, να βρούμε την ισορροπία και μπορεί να υπερβάλλουμε. Πρέπει να υπάρχει το σωστό περιβάλλον. Το σωστό περιβάλλον είναι μερικές φορές πολύ καλύτερο από το να υπάρξουν συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Ακούσαμε τις γενικές ε, παρατηρήσεις των συνεισηγητών, θα περιμένουμε την έκθεση και θα τα ξαναπούμε στις 20 Μαρτίου όπου θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης. Βλέπω ότι η συνεργασία μεταξύ των σκιωδών ε, και των εισηγητών είναι πολύ καλή και βρίσκω ότι και η συνεργασία μεταξύ των επιτροπών είναι εξαιρετική. Πολύ καλό παράδειγμα λοιπόν αυτό Μπορεί να έχουμε ομάδες επιτροπών, κλάστερες επιτροπών ε, στην ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί το ίδιο γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο άρα. Και αυτό το κλάστερ μεταξύ ΙΜΚΟ και ΙΤΡΕ είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι αξιόπιστο, ε, και ε, για μακροπρόθεσμη δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ τη φίλη Βίκη Φόρντ. Καλή επιτυχία στις επιτροπές μας. 20 Μαρτίου του 2017 είναι η επόμενη μας συνεδρίαση. 20 ναι, Μαρτίου θα κάνουμε την εξέταση και υποβολή προθεσμιών μέχρι ε, τις 22 Μαρτίου. Θα περιμένω με μεγάλη χαρά ε, το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ.